άρθρο 216 εδάφιο 3, η Επιτροπή, 211 ε, εδάφιο 3, η Επιτροπή η Συνταγματικών Υποθέσεων προβλέπει τα εξή. Το άρθρο 166, άρθρο 167, παράγραφος 1 και το άρθρο 195 εδάφιο 3 για την ονομαστική ψηφοφορία και για το άρθρο 6β εδάφια 2 και το 7 παραγραφή 3, 6 και 8 οι εκθέσεις μέσα στο πλαίσιο της άρσης ασυλίας δεν θα εφαρμόζονται. Αυτή η ερμηνεία θεωρείται ότι εγκρίνεται αν μέχρι την επόμενη περίοδο συνόδου δεν θα έχει υπάρξει ένσταση από μια κοινοβουλευτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτές. Το κείμενο της ερμηνείας αυτής θα το βρείτε στο Seance en Direct στην ιστοσελίδα. Ο κύριος Ιβαρη Πάνταρ από την 7η Απριλίου στην Εστονία διορίστηκε Υπουργό Γεωργίας. Ο κύριος Αρλέμ Ντεζίρ διορίστηκε την 9η ε, Απριλίου 2014 ως ε, ε, Υφυπουργό